πορεία, οπότε και ε, ούτως εγκρίνεται. Ε, δεύτερη ανακοίνωση. Σύμφωνα με το άρθρο 87α εδάφιο 6 του κανονισμού, ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής των Προέδρων Επιτροπών ε, μου διαβίβασε ότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις κατά της συστάσεως της Επιτροπής. Πρόκειται για την Επιτροπή Περιβάλλοντος για απόφαση ε, να μην προχωρήσουμε ε, σε ε, πρόταση για εφαρμοστικά μέτρα ενός κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αντικατάσταση, τροποποίηση προηγούμενου κανονισμού με βάση την εφαρμογή την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η πρόταση αυτή η σύσταση ε, θεωρείται εγκριθήσα εκτός αν ε, προβάλλουν έσταση 40 βουλευτές ή μια πολιτική ομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση ε, σε ψηφοφορία η σύσταση αυτή. Σε περίπτωση που θέλετε να διαβάσετε μπορείτε να τη βρείτε στο Seance on Direct και ε, μπορείτε να τη διαβάσετε. Αυτές ήταν οι δύο ανακοινώσεις μου και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα το σχέδιο συνθήκης του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Πνευματικής ή Διανοητικής Ιδιοκτησίας για ε, εξαιρέσεις στα δικαιώματα δημιουργίας.